οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές με ενημέρωσαν για αίτημα άρσης ασυλίας του κυρίου Νταν Νίκα. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού, το αίτημα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η κυρία Ρενάτε Βέμπερ φεύγει από την ομάδα του ΕΛΚ και από 17 Νοέμβρη 2014